Pan Przewodniczący! Please take your seats. Καθίστε παρακαλώ, συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος. It's just three minutes past three. Τρία, τρεις και τρία. Είναι λέει ο πρόεδρος, διότι πάει λάθος το ρολόι, πάει πίσω, άρα πρέπει να αρχίσουμε παραυτήκα. Ογκουάσαμ wznowienie... Στα πολωνικά. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας, είχαν σταματήσει 21η Δεκάτου του Ενεστώτος ναι, έτους. i teksty przyjęte z posiedzenia w 21 października. Τα πρακτικά τη συνεδρία τη 21 η Δεκάτου διατίθενται και σα ρωτώ αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις. Δεν βλέπω καμία ένσταση, επομένως εγκρίνονται τα πρακτικά εκείνα. Και θα προβώ τώρα εις κάποιες ανακοινώσεις. Πώς δεν λειτουργεί η μετάφραση, η διερμηνία. Λέει τρεις φορές ο πρόεδρος. Now it's okay. Α, τώρα δουλεύει. Σας ρώτησα για τα πρακτικά της 21ης Οκτωβρίου. Μήπως έχετε παρατηρήσεις. We accepted the minutes. Αφού δεν έχουμε ενστάσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Πριν αρχίσει η συζήτηση θα πρέπει να σας πω ότι στις 6 Νοεμβρίου ο ολέγ Κάσιν υπέστη επίθεση και ξυλοδαρμό. Πρόκειται για πράξη που θα πρέπει να καταδικαστεί. Θεωρούμε πάρα πολύ θετική την ταχύ αντίδραση των ρωσικών αρχών και το ότι ο πρόεδρος Μέντβεντεφ προσωπικά ασχολήθηκε με την ε, σύλληψη των ε, υπετίων. Στις 21 ε, Οκτωβρίου, για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, έγινε διαδήλωση της αντιπολίτευσης στην κεντρική πλατεία της Μόσχας. Θεωρούμε ότι πρόκειται για θετικό γεγονός και Αντιστοίχω και εμεί έχουμε ζητήσει περαιτέρω δημοκρατισμό τη χώρα και επομένω λέμε ότι οι ενέργειέ μα έχουν πιάσει τόπο. Τρίτον, πριν από κάποιε μέρε στην Βαγδάτη ε, σημειώθηκε επίθεση κατά χριστιανών οι οποίοι ασκούσαν τη λατρεία τους σε κάποια εκκλησία. Είχαμε θανάτους αλλά και τραυματίες. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προς πάντες να σεβαστούν την ε, ελευθερία της ε, θρησκευτική λατρείας και ότι θα πρέπει να καταδικαστεί κάθε βία η ενέργεια. Τέταρτον, στις 10 Δεκεμβρίου πρόκειται να λάβει μια χώρα, χώρα ε, μια εκδήλωση για την απονομή του βραβείου Νόμπελ. Οι δε κινεζικέ αρχέ έχουν προσπαθήσει να πιέσουν τα κράτη-μέλη να μην γίνει η εκδήλωση αυτή. Εμείς πάντως ε, πρεσβεύουμε το να τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα παντού και στην Κίνα. Κατά την εκδήλωση εκείνη θα εκπροσωπηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον επικεφαλή τη εκείνη την προσωπία τη Ένωση. Έχουμε τώρα κάτι διαδικαστικού χαρακτήρα. Θέλω τον λόγο κύριος Μπέλιγκερ τι φυσικέ καταστροφέ φοβερή ε, ε, ένταση χτύπησαν την περιοχή τη Ιταλία στο Βένετο πρόσφατα, Βιτσέντσα, Πάντοβα και Βερόνο. Ε, πρόκειται περί πλημμυρών καταστροφικών διαστάσεων που δημιούργησαν οι βροχοπτώσει περίπου 500.000 άτομα που επλήγησαν αυτόν τον τρόπο και εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ σε ζημιέ. Ε, τραγωδία γονάτισε όλε τι παραγωγικέ περιοχέ, τι μικρομεσαίε